Good morning, everybody. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε πολύ πιεσμένο χρονοδιάγραμμα σήμερα και πολύ λίγο χρόνο για ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να ξεκινήσω αμέσως, διότι βλέπω ότι Όλα τα μέλη που πρέπει να είναι εδώ είναι εδώ για το πρώτο τμήμα της ημερήσιας διάταξης. Να σας αναφέρω το γλωσσικό καθεστώς. Δυστυχώ δεν υπάρχει διερμηνία στα δανέζικα, μαλτέζικα, κροατικά και ιρλανδικά. Πρέπει να εγκρίνουμε και τις συστάσεις των συντονιστών για τον ορισμό εισηγητών. Ο κύριος Κορά από το EFTD είναι εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης για την αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων για την ε, ταξινόμηση των οχημάτων στην Πορτογαλία η Επιτροπή εγκρίνει τη σύσταση των συντονιστών. Εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Τώρα, για τις ε, κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις έχω στοιχεία για τρία θέματα για τον κανονισμό της 13ης Δεκεμβρίου του 2017 για την ε, προσθήκη της ε, Σρι Λάνκα, της Τρινιντάτ ε, και τον Πάκο και τη Δινησία... στο παράρτημα 1 του κανονισμού. Μετά από το αίτημα ένστασης από τρία μέρη της ΕΚΟΝ και της ΛΥΜΠΑ ξεκίνησε μια γραπτή διαδικασία στις 12 Ιανουαρίου και η πλειοψηφία των συντονιστών ΛΥΜΠΕ και ΕΚΟΝ αποφάσισαν ότι θα επιβάλλουν ένσταση και συμφώνησαν να συνεργαστούν στα αγγλικά μόνο και μέχρι τις 5 η ώρα στις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να δοθούν τα στοιχεία. Η κοινή συνεδρία θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου, 6.30 με 8. Πιθανή ψηφοφορία για το αίτημα της ένστασης ε, θα γίνει σήμερα για να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, ε, στην πρώτη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Στις 16 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε τον εκτελεστικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καθορίζει τους κανόνες για την εφαρμογή της οδηγια 1148 1148-2016 για τις περαιτέρω διευκρινήσεις για τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπεύθυνοι για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, για την ασφάλεια δικτύων και τα συστήματα πληροφορικής, η βασική πράξη που αφορά μέτρα για υψηλή ασφάλεια δικτύων και ε, συστημάτων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση. Στις 16 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε την εκτελεστική απόφαση που καθορίζει τον κατάλογο των συνοδευτικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλουν, ε, όσοι υποβάλλουν ε, αίτηση για, διάρκεια, για θεώρηση βραχίας παραμονής από την Αυστραλία και κάποιες άλλες χώρες. Τα έχετε όλα στο newsletter της Επιτροπής ΤΛΙΜΠΕ και επίσης υπάρχει και ηλεκτρονική ψηφοφορία σήμερα στις 11. Παρακαλώ φροντίστε λοιπόν να έχετε τις κάρτες σας. Και τώρα, αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για τα πρακτικά, εγκρίνουμε τα πρακτικά της 6ης ε, Νοεμβρίου και 8ης Δεκεμβρίου και περνάω απευθείας ε, στο πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξης. Θα ακούσουμε την παρουσίαση της έκθεσης της αντιπροσωπείας, του σχεδίου έκθεσης της αντιπροσωπείας της ε, αντιπροσωπείας της ΠΑΝΑ στη Μάλτα που έγινε 30 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου του 2017. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και τα μέλη της πρώην Επιτροπής ΠΑΝΑ που είναι εδώ για ανταλλαγή απόψεων και τον ε, Υπουργό Δικαιοσύνη της Μάλτας, τον κύριο Όουεν Μπονίτσι που ζήτησε να συμμετέχει στη συζήτηση και επίσης εξ όσων ενημερώνομαι είναι εδώ και τα παιδιά της ε, ε, της Κορουάνα, ε, της ε, εκλειπούσας Κορουάνα και τους καλωσορίζουμε εδώ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Η αποστολή αυτή ήταν συνέχεια της ε, απόφασης των συντονιστών και έγκρισης από τη διάσκεψη των Προέδρων η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ότι θα μπορούσε να πάει μια ad hoc αντιπροσωπεία 8 μελών, ένα από κάθε πολιτική ομάδα και κατά πάσα πιθανότητα από την Επιτροπή Πολιτικών ε, ε, Ελευθεριών και της Επιτροπής ε, ε, της ΑΤΧΟΚ για την ε, παρακολούθηση της νομιμοποίησης παρανόμενων εσόδων και της ευρωδιαφυγής. Θα δώσω το λόγο αμέσως στην Άννα Γκόμες ως πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για να μας πει τι διαπίστωσαν κατά την αποστολή. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να ζητήσω την κυρία Γκόμες να τηρήσει το όριο των 10 λεπτών και από εκεί και πέρα τα άλλα μέλη και συντονιστέ από δύο λεπτά θα είμαι πολύ αυστηρή με το χρόνο για να μπορέσουν όλοι να μιλήσουν σήμερα το πρωί. Κυρία Γκόμες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καταρχάς επιτρέψτε μου να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό. Αυτό ακριβώς θέλουμε, να συνεχίσουμε ε, τις συζητήσεις με τις αρχές και τους ενδιαφορομένους στη Μάλτα για να διευκρινίσουμε πολλά από τα θέματα τα οποία χρήζουν διευκρίνησης όπως ε, ε, θα διαπιστώσει οποιοδήποτε διαβάσει την έκθεση από την αποστολή. Η έκθεση είναι αρκετά περιγραφική ε, και εξηγεί τι ακριβώς βιώσαμε. Και να καλωσορίσω και τους τρεις γιους της εκλειπούσας κυρίας Ντάφνε Γκαρουάνα Γκαλίτσια και τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένειά σας. Η έκθεση, όπως σας είπα, ε, είναι αρκετά περιγραφική. Γνωρίζουμε το πλαίσιο, τι κάναμε, τι μας είπαν στη Μάλτα Βεβαίως ε, τα μέλη ήταν προετοιμασμένοι, ε, συνέλεξαν πληροφορίες, έθεσαν ερωτήσεις και πήραν απαντήσεις. Και αυτό το οποίο έχει σημασία στην έκθεση είναι το δεύτερο σκέλος, στο οποίο αναφέρουμε τα βασικά μας ε, πορίσματα, δεν θα σας τα διαβάσω τώρα, και κάνουμε και συστάσεις. Συστάσεις προς τις αρχές της Μάλτης, Μάλτας και συστάσεις προς τις ευρωπαϊκές αρχές, γιατί αυτό το οποίο ε, κάνουμε στη Μάλτα δεν αφορά μόνο τη Μάλτα, αφορά όλους εμάς, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και μας ε, επηρεάζει όλους υπό την έννοια ότι το ξέπλυμα χρώμα, χρήματος, η διαφθορά έχει ε, συνέπειες για όλους. Είναι θέμα λοιπόν γενικού ενδιαφέροντος και αφορά και την ασφάλειά μας θα μπορούσα να πω. Η δήλωσή μου αυτή τη στιγμή ε, θα ήταν ίσως πιο χρήσιμη αν σας εξηγήσω απλώς τα γεγονότα. Τι ακριβώς δηλαδή προέκυψε από όλες αυτές τις επαφές ε, που είχαμε στη Μάλτα. Πρώτον, υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ε, αναφέρονταν στα Panama Papers και ήταν βέβαιο ότι υπήρχαν και ε, εκθέσεις ε, της Μάλτας, ε, πολιτικά εκτεθειμένα άτομα στην κυβέρνηση και που παρέμειναν στην κυβέρνηση. Ο ένας είναι υπουργό, ο κύριος Μίτσι και ο άλλος βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι γεγονός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται διεφθαρμένοι σε όλη τη Μάλτα ε, υπάρχουν εκθέσεις οι οποίες έχουν διαρρεύσει ε, στον τύπο και δεν ε, ανελήφθη καμία δράση, τουλάχιστον από πλευράς αστυνομίας. Η αστυνομία και ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έλαβαν υπόψη τους αυτές τις εκθέσεις. Κάποιες από αυτές έχουν δημοσιοποιηθεί και ε, παρόλα αυτά υπάρχουν πέντε ε, δικαστικές έρευνες ε, εν εξελίξη και εάν ολοκληρωθούν υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να οδηγήσουν σε κάποια αστυνομική δράση. Και σε αυτές τις πέντε δικαστικές έρευνες η μία έχει διακοπεί, την έχει μπλοκάρει η κυβέρνηση και αφορά τα πολιτικά εκτεθειμένα αυτά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στα Panama Papers ε, και στις εκθέσεις ε, αυτές. Επίσης ένα άλλο πάρα πολύ τραγικό γεγονός είναι το γεγονός ότι η Ντάφνε Καρούανα Γκάλη δολοφονήθηκε και ήταν και ε, δημοσιογράφος, blogger η οποία εξέθετε τη διαφθορά και κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους ε, ε, που ε, είναι εκτεθειμένοι στα Panama Papers. Πριν φύγουμε για τη Μάλτα, δύο μέρες πιο συγκεκριμένα πριν, η ύποπτη για την δολοφονία της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια συνελήφθησαν και ε, είναι υποκράτηση αυτή τη στιγμή και θα μπορέσουν ίσως να διευκρινίσουν και ποιος ε, διέταξε αυτή την δολοφονία γιατί είναι σαφές ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται από αυτή, ε, πίσω από αυτή τη βομβιστική επίθεση και θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι και για ποιο σκοπό έγινε αυτή η βομβιστική επίθεση και ε, η οικογένεια διαμαρτύρεται ότι δεν ενημερώθηκαν, δεν τους ενημέρωσαν ότι ε, συνελήφθησαν οι φερόμενοι δράστες ε, και υπάρχουν και κάποια στοιχεία που αφορά την ε, ε, σχέση μεταξύ οικογένειας και ανακριτικών αρχών ε, και δεν υπήρχε αυτή η επικοινωνία. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι ο πρώην Μαλτέζος Επίτροπος, ο κύριος Τζον Ντάλι, ο οποίος υποχρώθηκε σε παρέτησε για πάρα πολύ σοβαρές κατηγορίες και ισχυρισμούς ε, διαφθοράς και δωροδοκίας και παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια πάρα πολύ σοβαρή και αναλυτική έρευνα της Όλαφ ε, και από τις Μαλτέζικες αρχές ε, οικονομικού εγκλήματος υπήρχε και σχετική έκθεση, δεν έγινε ποτέ τίποτα, δεν τον άγγιξε κανείς και μάλιστα είναι και σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολύ συχνά στη Μάλτα ακούμε κάποιες ερμηνείες ότι ε, όλα αυτά είναι ανταλλάγματα, υπάρχει μια πολιτική διένεξη μεταξύ των δύο βασικών ε, ε, κυρίαρχων κομμάτων. Αλλά το άτομο αυτό ανήκε στο Εθνικό Κόμμα, στο Nationalist Party και έγινε σύμβουλος του αντιπάλου κόμματος. Πρέπει να δούμε λοιπόν γιατί δεν αναλήφθη καμία δράση και πρέπει να δούμε τι σχέση υπάρχει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο το οποίο είναι γεγονό. Ο κύριο Φέρη, ένα whistleblower πληροφοριοδότη που συναντήσαμε, ε, ήταν αντικείμενο μιας επίσημης αστυνομικής έρευνας, ε, ε, δεν υπήρξε κάποια δίωξη στη συνέχεια, αλλά Πέρασαν δύο μήνες και παρά το γεγονός ότι ε, πιέσαμε και τον Πρωθυπουργό και την αστυνομία ότι χρειάζεται προστασία και ο ίδιος και η οικογένειά του. Έχουν περάσει δύο μήνες ε, και δεν έχει ακόμα λάβει καθεστώς ε, whistleblower και του ζητάνε να δώσει πρώτα τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του στην κυβέρνηση πριν του δώσουν τέτοιο καθεστώς. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι υπάρχει ε, πώληση διαβατηρίων εθνικότητας Μάλτα, υπάρχει ένα σχετικό πρόγραμμα, υπάρχουν ε, αποδείξεις ότι είναι μια πολύ διεφθαρμένη υπόθεση, υπάρχουν άνθρωποι που πουλούν αυτά τα διαβατήρια, υπάρχει και, και κάποιες αποκαλύψεις στα Panama Papers επ' αυτού και ζητήσαμε ε, να έχουμε ένα κατάλογο των ατόμων που έχουν λάβει αυτό το ειδικό καθεστώς ε, συνήθως υπάρχει ένα κατάλογος ανθρώπων που ε, λαμβάνουν ηθαγένεια μέσω αυτής της διαδικασίας και δημοσιοποιείται. Γιατί δεν υπάρχει λοιπόν δημόσιος κατάλογος, ε, γιατί είναι όλα αυτά και καλυμμένα και δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι υπάρχει μια πολύ ανησυχητική σχέση μεταξύ της ε, Τράπεζας Πιλάτες, η οποία βρίσκεται στο κέντρο όλης αυτής της έρευνας ε, και του κυρίου Μπατζάνη. Θα πρέπει να σας πω ότι χθε το βράδυ κάποιος από εμά ε, τις πρώτες πρωινές ώρες ε, λάβαμε μία ενημέρωση από την τράπεζα. δεν είχα χρόνο να το διατρέξω, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα το αναλύσουν και τα μέλη της Επιτροπής. Το γεγονός είναι ότι αναγνωρίζετε ότι δεν είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας και είναι ανησυχητικές αυτές οι σχέσεις ε, και πρέπει να ανησυχεί κυρίως και την κυβέρνηση της Μάλτας. Και κάτι ακόμα. Υπάρχει και η οδηγία υπαριθμών 4 της καταπολέμησης της νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων που θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο και ακόμα δεν εφαρμόζεται στη Μάλτα. Θα μπορούσα εδώ να αναφερθώ και σε πολλά άλλα πράγματα, πολλές ε, υποθέσεις ε, δωροδοκίας, ε, ξένες δικαιοδοσίες οι οποίες κινούνται κατά Μαλτέζων δημοσιογράφων για να τους φημώσουν. Ε, θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε ερωτήσεις αν έχουμε χρόνο, κυρίως προς τον Υπουργό, ο οποίος ε, ε, είναι πολύ σημαντικό ότι ήρθε εδώ να συζητήσει μαζί μας. Δεν ξέρω αν έχω ερωτήσεις τώρα. Αν έχουμε τη δυνατότητα θα θέσω αυτές τις ερωτήσεις και σχετίζονται και με όλα αυτά τα στοιχεία και με τις απαντήσεις τις οποίες πρέπει να λάβουμε. Μία ερώτηση μόνο να κάνω αυτή τη στιγμή. Η Ντάφνη Καροάνα Γκαλίτσια δημοσίευσε μία σειρά μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21 Μαΐου πέρσι που αποδείκνυαν ότι ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός και άλλα μέλη της κυβέρνησης μαζί με ε, μέλη της επιχείρησης ε, που ασχολείται με την πώληση των διαβατηρίων. απειλούσαν να ε, Υποβάλλουν μήνυση και να ζητούν ε, χρηματική αποζημίωση ε, κατά της Δάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια. Είναι περίεργο να υπάρχει σχέση των Μαλτέζικων αρχών ε, με αυτή την επιχείρηση και να απειλούν έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο και blogger. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ερώτηση που θα ήθελα να θέσω στον Υπουργό. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι στα 10 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου θα μπορούσα να τις θέσω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία Κόμες. Και τώρα έχουμε να εκπληρώσουμε το αδύνατο αυτό καθήκον του να οργανώσουμε τη συζήτηση σε μία ώρα. Έχω τόσο πολλούς ομιλητές. Να σας πω λοιπόν πώς θα κινηθούμε. Θα ακούσουμε καταρχάς τους συντονιστές, ένα γύρο συντονιστών από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και από την Επιτροπή ΠΑΝΑ. Στη συνέχεια θα περάσουμε στα μέλη της Επιτροπής, της Αποστολής, συγγνώμη, και μετά στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Και θα σας ζητήσω πραγματικά να περιοριστείτε σε δύο λεπτά, γιατί ιδάλω δεν θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο καν τα μέλη. Ό,τι και να κάνουμε, η κυρία Μέτσολα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και να ξεκινήσω ευχαριστώντα την προσωπία που έκανε τη δουλειά τη για την αποφασιστικότητα και την εντελέχεια τη. υπό συνθήκε δύσκολε να το ξεκαθαρίσω ευθύ εξ αρχής, ότι η σαπίλα που αποκαλύφθηκε στην αποσταλή αυτή δεν είναι αντιπροσωπευτική της Μάλτας και του Γκόζο, αλλά καταδεικνύει πόσο κατεπηγόντως χρειάζεται ανάληψη δράσης σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους, την ε, αστυνομία. Συναντήθηκαν με όλους τα μέλη της αποστολής και νομίζω ότι σχημάτισαν μια πολύ σωστή εικόνα. Όχι, όχι ότι χρειάζονταν η αποστολή του Κοινοβουλίου να μα ε, πει ότι ήταν απαράδεκτο το ότι η αστυνομία την αντέδρασε σε τέτοιε κατηγορίε δωροδοκία, ε, ξεπλήματο δρομικού χρήματο, για το γεγονό, για παράδειγμα, επίση ότι οι πληροφοριδότε δεν μπορούν να τεθούν στο στόχαστρο και να, προσ... να προστατεύονται, ή ότι, για παράδειγμα, οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν την ελευθερία να γράφουν. Όλα αυτά είναι αυτονόητα. Ο Πρωθυπουργό μα ε, χαμογέλασε και δεν έδωσε άλλη προσοχή στην αποστολή και σήμερα, αυτή την εβδομάδα, 100 ε, ημέρες μετά την τηλεφωνία της Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια, βγήκαν και είπαν ότι όλα πάνε καλά στη Μάλτα και δημοσιεύτηκαν αυτά στις εφημερίδες και ότι α, ας, έγραφε αυτή ό,τι ήθελα. Απάντησαν λοιπόν οι ηγητής ότι πώς είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά τη στιγμή που δολοφονήθηκε για αυτά που έγραψε. Ο μηχανισμός λοιπόν ε, του, της κυβέρνησης ε, στράφηκαν κατά ημών και θα συνεχίσουν. Αλλά δεν πρόκειται να ε, υποχωρήσουμε έναντι αυτής της Όχι, προασπιζόμαστε και υπερασπιζόμαστε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε γιατί η Μάλτα πρέπει να είναι μια χώρα όπου υπάρχει σωστό, σωστή εφαρμογή του δικαίου και όπου οι δημοσιογράφοι μπορούν να γράφουν ε, χωρίς να εκτελούνται. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί το κράτος δικαίου και η δουλειά μας είναι εδώ να δείξουμε σε όλους και όσου, όλους όσοι παρακολουθούνται ότι η Μάλτα, δεν μπορεί να, η Μάλτα και η Μαλτάζικη κοινωνία δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από τους απαταιώνους αυτούς και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μέτσολα, η κυρία Σίπελ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε τα Pana Papers και τα Paradise Papers. Γιατί? Γιατί οι δημοσιογράφοι έκαναν καλά τη δουλειά τους και γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε την Επιτροπή πάνω εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο και ελπίζω να ξεκινήσει και άλλη μια τέτοια Επιτροπή μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα. Το περιεχόμενο δε των ε, Pana Papers και των ε, Paradise Papers αυτό ήταν που μας οδήγησε στην αποστολή στη Μαλτά. Όχι, όχι, εκτέλεση μιας δημοσιογράφου που ήταν αυτή που μας ανάγκασε να κάνουμε μια αποστολή στη Μάλτα και εδώ έχουμε δύο στοιχεία τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουμε. Η πρώτη ερώτηση που προκύπτει είναι το θέμα τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Να ελέγξουμε κατά πόσο στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για κάτι συστηματικό το οποίο συμβαίνει πει Πέρα από αυτό, φυσικά, του ποιου, το ερώτημα του ποιο έδωσε την εντολή για την εκτέλεση της δημοσιογράφου. Όλα αυτά χρήζουν περαιτέρω έρευνας. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει. Και θα πρέπει να ελέγξουμε όλους αυτούς, να διερευνήσουμε όλους αυτούς τους τομείς. Και γι' αυτό λοιπόν και ξεκινάει αυτή η ειδική επιτροπή στο Κοινοβούλιο. Εκ παραλλήλου, εκτιμώ το γεγονό ότι ο Υπουργό Δικαιοσύνη τη Μάλτα είναι σήμερα μαζί μα και είμαι πεπισμένη ότι θα έχει και δικέ του ιδέε να προτείνει για το πώ θα αντιδράσει στην έκταση της αποστολής και σε όλα τα οποία, αυτά τα οποία περιέχει. Αλλά θα ήθελα να κάνω και κάποιες ερωτήσεις. Αν δεν μπορείτε να τις απαντήσετε λόγω χρονικών περιορισμών, ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε και κάποιες απαντήσει γραπτά εκ των υστέρων. Δύο ερωτήσει λοιπόν έχω μόνο να απευθύνω. Η πρώτη είναι η εξή, ότι ο Γενικό Εισαγγελέα που εξετάζεται τακτικά από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πείτε μας, ποια ήταν η πρόσφατη αξιολόγηση λοιπόν του Συμβουλίου της Ευρώπης για το θέμα αυτό. Και δεύτερη ερώτηση, το σύστημα ερευνών σας για την ε, λειτουργία της εισαγγελία και του δικαστικού σώματος, πώς λειτουργεί στην Μάλτα, ερευνάτε όσα έλεγε και έγραφε η Ντάφνε ε, Καρουάνα Γκαλίτσια ε, στα, Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Σάιμον από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες από την Επιτροπή Πανά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να βάλετε και τα ακουστικά σας, παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία για την έκθεση που μας υπέβαλα και εκ νέου είμαστε αντιμετωποί με πολλά ερωτηματικά για ένα κρατός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι και η πρώτη φορά που στα πλαίσια των ερευνών της Επιτροπής ΠΑΝΑ και της προηγούμενης Επιτροπής ε, τάξε 1 και τάξε 2 είμαστε αντιμέτωποι λοιπόν με ένα κράτος μέλος όπου λαμβάνουν χώρα ε, διαδικασίες οι οποίες χρήζουν ανταλλαχέστερης ε, μελέτης. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ως Κοινοβούλιο να θέσουμε ένα μήνυμα. Τώρα σε ό,τι αφορά δηλαδή τις εργασίες της Επιτροπής Πάνα η οποία ολοκληρώθηκε να συνεχιστεί, να συνεχιστούν οι εργασίες της αυτές και να ασχοληθεί με τα ερωτήματα που έθεσε η κυρία Γκόμε για τη Μάλτα, αλλά και με άλλα ερωτήματα για άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε καθαρά. Θα πρέπει να είμαστε σαφεί και ξεκάθαροι και δικαίοι. Και θα πρέπει τα μέτρα που θα θέσουμε και τα σταθμά να φροντίσουμε να ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά να ισχύουν και τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν και για τρίτε χώρες και που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σα υπενθυμίσω ότι από τον κατάλογο φορολογικών παραδείσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε διαγράψει διάφορες χώρες. Κοιτώντας λοιπόν τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση σε ό,τι αφορά τη Μάλτα καθώς και σε ό,τι αφορά και τις άλλες κατηγορούμενες χώρες, τι διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει στο Κοινοβούλιο να ελέγξουμε επακριβώς κατά πόσον στέκουν ε, οι αιτιάσεις και οι κατηγορίες και που από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Αλλά καταρχάς χρειάζεται αυτή η πρώτη έρευνα πρωτού να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από το ECR. Ο κύριος Λούκε, ο συντονιστής της Επιτροπής έπανα να Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και την αντιπροσωπεία η οποία μετέβη ε, στη Μάλτα. Θα πρέπει όμως να θέσουμε και το ερώτημα τι θα συμβεί όταν ε, το ε, Κοινοβούλιο, τι θα συνέβαινε άμα το Κοινοβούλιο δεν απέστελε μια τέτοια αποστολή. Τότε ποιος θα ασχολιόταν ούτως ώστε να λύσει τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην Μάλτα. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο συγκεκριμένο αλλά πρόκειται για διαρθρωτικές ε, δυσκολίες που έχει ε, η Μάλτα ε, βλέπουμε ότι οι δίωξη, οι διοκτικές αρχές είναι πολύ αργά, δεν είναι αξιόπιστες, υπάρχει τάση για νεποτισμό και αδιαφάνεια. Έχουμε πράγματα, τα οποία, φαινόμενα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατικότητα μιας χώρας και βλέπουμε για παράδειγμα ότι υπάρχει μια αποδοχή ε, για ε, πώληση υπηκοότητας ή αγοράς ψήφων Όλα αυτά λοιπόν είναι δυσκολίες ενός κράτους ε, μέλους που πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να ε, αναλάβει ε, μία δράση τέτοια διότι η Κομισιόν είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τις συνθήκες και θα πρέπει να διασφαλίσει ότι γίνονται πρόοδοι. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο σχετικά με αυτό το έλλειμμα το, οποίο το οποίο είσαμε στη Μάλτα, θα το παρακολουθήσουμε και θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα ελλείμματα. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο έργο για το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, ούτω ώστε η δολοφονία της Δάφνης ε, αλλά ε, και τα λάθη τα οποία παρατηρήθηκαν, όχι απλά να παρατηρηθούν και να μπουν σε ένα φάκελο, αλλά στη συνέχεια να βρεθούν και λύσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ε, Λίμπε. Άλντε, η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να ε, καλωσορίσω τα παιδιά της ε, κυρίας Γκαλίτσια όταν ε, διάβασα την αναφορά πραγματικά σοκαρίστηκα, ακούσαμε για διαφθορά, αλλά όταν είδα τις λεπτομέρειες σκέφτηκα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά είναι σοβαρό και περιγράφει πρακτικές οι οποίες ε, προφανώς είναι τόσο σκοτεινές ε, που κάποιος πίστεψε ότι μπορεί να σκοτώσει ακόμα για όλο αυτό. και θα πρέπει να... και προσπάθησε να το καλύψει. Ο κύριος Μόσκα τα σε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέλο του οποίου ήταν κάποτε. Και αυτό είναι ιδιαίτερα στενόχωρο, διότι το να απορρίπτει το Κοινοβούλιο σημαίνει ότι απορρίπτει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι παρακολουθούν Ταυτόχρονα όμως ε, είναι λάθος συμπεριφορά διότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα πολύ σημαντικό ε, ρόλο στο να ξεκαθαρίσει όλη αυτή την υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο δυνατή όσο ο πιο αδύναμος της Κρήκος και φαίνεται ότι η Μάλτα γίνεται αδύναμος Κρήκος. Τι, τι σημαίνει όλο αυτό με την αστυνομική και με τη συνεργασία των δικωτικών αρχών και τη συνεργασία με την Europol. Αν δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις πληροφορίες που δίνονται στο σύστημα, τότε πώς είναι δυνατόν να διασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια και την νομοθεσία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ε, πρέπει ε, να εργαστούμε με βάση την, υπό, την, με βάση την υπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες κάποια ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να θέσω προς την Κομισιόν αλλά και τον Υπουργό. Η δολοφονία της κυρίας Γκαλίτσια ήταν ε, πριν από ακριβώς τρεις μήνες. Ε, τι πρόοδος υπάρχει όσον αφορά την έρευνα και θα μπορούσε να μου εξηγήσει κανείς αν η σύλληψη των τριών έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη. Διότι δεν είμαι αστυνομικός, αλλά όταν διαβάζω όλο αυτό στις ε, εφημερίδες μου φαίνεται ότι όλο αυτό είναι ένα πανηγύρι. ήταν πολιτική δολοφονία δεν ήταν κάποιο που ήθελε να τη κλέψει την τσάντα. Ε, ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι γίνεται λοιπόν ε, με την έρευνα. Ε, τώρα όσον αφορά τις χρυσές θεωρήσεις είναι κάτι ε, στο οποίο μας ε, ενημέρωσε η Μάλτα. Υπάρχουν παρόμοια σχέδια και σε άλλα κράτη-μέλη, ε, όμως είναι καιρός πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον να καθαρίσει αυτό το θέμα, όπως επίσης και τις άδειες διαμονές μεταναστών και προσφύγων. Πόσα χρήματα επίσης ήρθαν στον κριτικό κορβανά από όλα αυτά. Διότι δεν πρόκειται για ηλικιωμένε ε, γιαγιάδε από τη Ρωσία. Πολύ φοβάμαι ότι ε, φέρνουμε ε, χρήματα από παράνομες δραστηριότητες. Και τέλος, προσπαθή, θελήσατε να ακυρώσετε την αιτήσια αναφορά παρανομίας, τη διαφθοράς. Θα ήθελα λοιπόν από την Επιτροπή πώς πρόκειται να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο όταν δεν το κάνουμε, χρησιμοποιώντας μια αιτήσια αναφορά. Η κυρία Παγκάζα ως συντονίστρια ε, της ΑΛΔΕ από την Επιτροπή ΠΑΝΑ. Σας παρακαλώ, ε, κρατήστε το χρονοδιάγραμμα των δύο λεπτών. Ε, δεν θέλουμε να στερήσουμε το χρόνο από του συναδέλφου. Παρακαλώ. Ναι, η κυρία Παγκαθαρό Ουρτουνδία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Αποστολής για τα στοιχεία που μας έδωσαν μας ε, τρομοκράτησε η όλη κατάσταση και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θεωρείτε ότι ε, το αίτημα πληροφοριών για αυτό τον κατάλογο που παίρνουν αυτές τις χρυσές ε, θεωρήσεις θα γνωστοποιηθεί. Ε, μπορεί να μην έχουμε αρμοδιότητα να είμαστε θεματοφύλακες των συνθήκων, αλλά έχουμε πολιτική αρμοδιότητα, γιατί είμαστε κοινοβούλιο. Και εμείς πιστεύω ότι έχουμε την ε, πολιτική και ηθική ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν και συνέβησαν με την Τάφνε καρούανα να προχωρήσουμε και δεν μπορούμε να αφήσουμε την αρμοδιότητά μας ε, να είναι απλώς κενά λόγια τα οποία θα χαθούν σε ένα σιρτάρι. Πρέπει να ε, παρακολουθήσουμε την υπόθεση και να υπάρξει μια συνέχεια. Ε, να δούμε τι έχουμε ερευνήσει στην Ειδική Επιτροπή, γιατί είναι υποχρεωτικό να γίνει, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η δουλειά μας, γιατί υπάρχουν διαρθρωτικά ζητήματα, γιατί το άρθρο 2 της συνθήκης ε, ε, σίγουρα δεν εφαρμόζεται σωστά στη Μάλτα και θα ήθελα να ευχαριστήσω και θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτοί που ήταν στην αποστολή στη Μάλτα πιστεύουν ότι θα λάβουμε επαρκείς πληροφορίες. Ευχαριστούμε την κυρία Πακαθάρα Ουρτουντούα. Συντονιστής των πρατήσεων τώρα, ο κύριος Γκίγκολτ. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συνεργασία. Το τελευταίο έτος να ευχαριστήσω και τον ε, Υπουργό, να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως και τους γιους της Δάφνη Καλήσια που βρίσκονται εδώ σήμερα. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να βρούμε μία ευκαιρία να πάρουν και αυτό το λόγο, γιατί νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να πάρουν και αυτοί το λόγο να μιλήσουν και να πούν τι θέλουν να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν. Αυτό που κατέστησε σαφέ στην τελευταία επίσκεψη είναι ότι μάθαμε ότι το θέμα δεν είναι μόνο το ξέπλυμα χρήματος και οι αποκαλύψει σε των Pana Papers. Υπάρχει μία νοοτροπία τιμωρησίας συστημική και ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχουν υψηλού επίπεδου περιπτώσεις διαφθοράς, υποθέσεις διαφθοράς που να οδήγησαν σε επίσημες ε, έρευνες, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ε, τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί λοιπόν η ηλέκτρογας ε, η περίπτωση αυτή δεν ερευνήθηκε σωστά, γιατί η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων δεν ερευνήθηκε κανονικά, σωστά. Γιατί υπάρχει ένα κράτος μέλος όπου άμα ο υπεύθυνο δικαιοσύνη αναφέρει ότι υπάρχει επιδείνωση του κράτου δικαίου. Αυτά είναι ανησυχητικά. Επίση υπάρχουν σημάδια επιρροή του εκλογικού σώματο. με εξαγορά ψήφων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Θα πρέπει να τα πάρουμε όλα αυτά πολύ σε σοβαρά σε ό,τι αφορά και το NXBT, όπου ενημερωθήκαμε ότι δεν εφαρμόστηκε το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν υπήρξε ιδέουσα επιμέλεια και παρόλα αυτά δεν ακολούθησε καμία έρευνα. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και γι' αυτό λοιπόν καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τη δουλειά της, να συζητήσει μαζί μας και ελπίζω και το Κοινοβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες του. Μία ερώτηση προς τον Υπουργό. Μπορείτε να ενημερώσετε τον Κοινοβούλιο για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τις αιτιάσεις αυτές. Ενημερώστε παρακαλώ το Κοινοβούλιο για το τι πληροφορίες χορηγήσατε εγγράφος και μπορείτε να απαντήσετε επίσης γραπτά και στην εκθεσή μας. Αυτό θα μας βοηθούσε ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την πρότασή σας να ακούσουμε και να πούν δύο λόγια και η γη της κυρίας Ντάφνη Καρουάνα, αλλά να πω ότι μιας και είχατε και εσείς ε, συμμετείχατε στην αποστολή, είχατε δύο λεπτά λοιπόν ε, χρονομιλίας ως μέλη της αποστολής, μπορείτε να τα δώσετε στους γιους της Ντάφνη Καρουάνα. Βεβαίως, λέει ο κύριος Κίγκολτ, με χαρά. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τους συντονιστές. Η κυρία Κάπελ από το ΙΝΕΦΕ. Μίλησαν λοιπόν όλοι οι συντονιστέ και τώρα να περάσουμε στα μέλη της αποστολής. Ο κύριος Κάζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συναδέλφους και να τους ευχαριστήσω για την επαγγελματικότητα, τον επαγγελματικό χαρακτήρα της έκθεσης αυτής. Είναι σαφής η έκθεση και είναι σαφή και τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Η βασική ανησυχία προφανώς είναι ότι άτομα στους υψηλούς κύκλους της κυβέρνησης ε, θεωρούνται, θεωρείται ότι εμπλέκονται ενδεχομένω σε εγκληματικέ δραστηριότητε και παραμένουν ε, ατιμόρυτε και δεν ερευνώνται καν σήμερα. Η τράπεζα που χρησιμοποιήθηκε για την νομιμοποίηση παρανομών εσόδων εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Και έχουμε και την ε, υπηρεσία την σχετική δικαιοσύνη τη Μάλτα, η οποία ζητά να ερευνηθούν τα περιστατικά αυτά και παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία συνέχεια. Και η εκτέλεση προφανώ τη Ντάφνε Καρουάνα, η τράπεζα πιλάτε εξακολουθεί να έχει ε, άδεια για να λειτουργεί. Είναι εξαιρετική, παίρνει ακόμα κρατικές προμήθειες και σήμερα είναι εδώ πέρα μαζί μας ε, ο κ. Μπονίτση. Τι θα μας πει όμως. Ε, θα μας πει ότι η κυβέρνηση του πέρασε νομοθεσία για τους ε, πληροφοριοδότες. Δεν θα μας πει όμως ότι προστατεύουν μόνο οι πληροφοριοδότες που συμφέρουν την κυβέρνησή του. Θα μας πει ότι πέρασε νομοθεσία για την διαφθορά. Αυτό που δεν θα μας πει όμως είναι ότι υπάρχουν πολιτικοί όμοιροι του ΕΦΑΙΟ και της αστυνομίας προκειμένου να μην ε, διώκονται ποτέ οι συναδελφοί τους. Θα μας πει ότι πέρασε νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης. Ε, δεν θα μας πει όμως ότι τα... Ε, οι λογαριασμοί της Ντάφνη Κορουάνα παραμένουν παγωμένοι και ήταν παγωμένοι τη στιγμή της εκτέλεσής της λόγω έρευνας για αυτά που έγραφε. Δεν θα μας πει για παράδειγμα ότι ο Πρωθυπουργό έκανε καταγγελία για να μην ενερευνηθούν οι συνεργάτες του. Θα προσπαθεί λοιπόν να τα παρουσιάσει όλα αυτά ως μια επίθεση για, κατά της Μάλτας. Η επίθεση όμως είναι υπέρ της Μάλτας, κατά της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γκραπίνη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και γιατί είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή την αποστολή στη Μάλτα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τα συμπεράσματα, γιατί οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν ήδη ε, σε αρκετά πράγματα. Καταρχάς ε, πιστεύω ότι η περίοδος ε, που έχουμε για την ανάλυση είναι πολύ μικρή. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ με αυτή την έκθεση και αυτή την ανάλυση. Δεν νομίζω ότι καταφέραμε να συναντήσουμε όλους τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην ανάλυση μας για την κατάσταση της Μάλτας. Για παράδειγμα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με όλους τους εκπροσώπου της κοινωνία των πολιτών ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν λάβαμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας από το Γενικό Εισαγγελέα. Ε, εγώ τον ρώτησα προσωπικά γιατί η των μεσων μαζικης ενημερωσης δεν λαβαμε απαντησεις στις ερωτησει μας απο το γενικο εισαγγελεα ε εγω τον ρωτησα προσωπικα γιατι η ερευνα για τη δολοφονία της ε, Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια καθυστερεί τόσο πολύ και δεν μου απάντησε. Όταν συναντήσαμε τον τύπο δεν λάβαμε απαντήσεις ε, ε, στην ερώτηση του κατά πόσον ε, πήραν τις πλήρεις εκθέσεις όταν ε, έγραψαν τα άρθρα για τα οικονομικά σκάνδαλα. Ε, δεν λάβαμε λοιπόν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και πρέπει να γίνει και σωστός επιμερισμός. Συναντήσαμε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Συναντήσαμε έναν κύριο Μιχαήλ Ντεγκούλιο που είναι και σύμβουλος του Εθνικού Κόμματος. Δεν ξέρω πόσο ε, σωστό είναι αυτό από δεντολογική σκοπιά. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα δικαιώματα των πολιτών και τις ζωές των πολιτών, γιατί εδώ έχει δολοφονηθεί μια δημοσιογράφος και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. τα δικαιώματα των πολιτών ε, για ελεύθερη έκφραση θα πρέπει να προστατεύονται και να γίνονται σεβαστά με καλύτερο τρόπο. Ε, μας εξέπληξε ότι συναντήσαμε τον κύριο Όστιν Γκάτ, ο οποίος ήταν πρώην ε, υπουργό και ήταν εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης. Είχε μπλακεί και σε ένα σκάνδαλο για πετρέλαια, υπήρχε λόγος για λογαριασμούς στην Ελβετία και ούτω καθεξής. Θα πρέπει λοιπόν να μην σκεφτόμαστε πού ανήκουν πολιτικά όλα αυτοί, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε τα δικαιώματα και τι ελευθερίε των ανθρώπων τη Μάλτα. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο για να λύσουμε την κατάσταση. Ο κ. Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά την κυρία Γκόμες και όλα τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής στη Μάλτα. Ε, χάρη στη λαμπρή μας συνεργασία εξεπλάγει και εγώ από τα αποτελέσματα αυτής της αποστολής, αλλά θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό δεν είναι πρόβλημα της Μάλτας, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Εάν δεν το ε, αντιληφθούμε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη Μάλτα. Στη Μάλτα υπάρχουν πάρα πολύ ε, σκοτεινές διαδικασίες και θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουν και να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Παραδείγματο χάρη, η Τράπεζα Πιλάτους Πώς μπορούμε να δεχθούμε ότι η τράπεζα έχει 130 ενδιαφερομένους μετόχους μόνο και από την άλλη είναι αδιανόητα τα ποσά των χρημάτων που βρίσκονται στις κατεθέσεις τους. Είναι κάτι το οποίο είναι κατανόητο, δεν μπορούμε να το δεχτούμε έτσι αυλεπή, όπως είπα. Ε, κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω, γιατί τα μέλη της αποστολής ήδη τα είπαν όλα, είναι κάτι που αφορά την κυρία Μαρία Φίμωβα που είναι whistleblower και μας μίλησε ε, μέσω Skype. Υπάρχει ένταλμα διοξίστης στην Κύπρο, θέματα. Και δεν ξέρω αν αυτά σχετίζονται με το γεγονός ότι είναι πληροφοριοδότης. Εγώ με την κυρία Γκόμε, ε, ήδη έχουμε συντάξει μια επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου για να μας πει δύο λόγια για αυτού τους ισχυρισμού ε, και γιατί ε, υπάρχει διεθνές και ευρωπαϊκό ένταλμα κατά της κυρίας αυτής. Και επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τους γιους της κυρίας της Καρουάνα Γκαλίτσια και να τους εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα να περάσουμε στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής ε, που θέλουν να λάβουν το λόγο. Έχω τρία μέλη που έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Μπέκερ, η κυρία Φαγιόν και ο κύριος Ζάμι. Κλείνει ο κατάλογος των αγοριτών. Κύριε Μπέκερ, παρακαλώ, προσπαθήστε να είστε σύντομος. Ε, ούτε δύο λεπτά, βοηθήστε με παρακαλώ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Να ευχαριστήσω τη συνάδελφο την Ανάγκο, μέσα ε, για την έκθεσή της για την αποστολή στη Μάλτα. Τα βασικά συμπεράσματα στα οποία μπορούμε να καταλήξουμε σήμερα, όχι μόνο όσον αφορά το κράτος δικαίου, το ξέπλυμα χρήματος, ε, αλλά και ε, μια απίστευτη ιστορία υπόπτων δολοφονίας με ένα πολύ σοβαρό ε, υπόβαθρο ε, διαφθοράς ε, ανθρώπων που προστατεύονται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές σε υψηλά ιστάμενες θέσεις της κυβέρνησης. Και θα ήθελα καταρχάς να διευκρινίσω ότι ο λαός της Μάλτας δεν αξίζει αυτή την εικόνα ανά τον κόσμο. Οι υπεύθυνοι κυβερνητικοί ηθήνοντες θα έπρεπε να είχαν παρετηθεί εδώ και μήνες. Πρέπει να υποστηρίξουμε το λαό της Μάλτας και να συνεχίσουμε να διώκουμε τα διεφθαρμένα ε, μέλη που είναι εγκληματία σε οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκονται, ακόμα και στην κυβέρνηση της Μάλτας. Είναι απαράδεκτο λοιπόν εγκληματικά στοιχεία να ζητούν στη Μάλτα ακόμα και η σύλληψη του Ευρωβουλευτή του Νταβίτ Κάσα ο υπαριθμόν ένα άνθρωπος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος ε, ε, δίνει μάχη για να βρεθούν αυτές οι υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης, ακόμα και αυτόν τον βίαιο θάνατο ε, στη Μάλτα. Όλα οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι στη Μάλτη από εδώ, ακόμα και εσείς ε, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, ε, ε, να ξέρετε ότι εμείς υποστηρίζουμε πλήρως τον Νταβίτ Κάσα και δεν θα τα καταφέρετε. Θα πρέπει οι άνθρωποι στη Μάλτα να υψώσουν το ενόστημά τους εναντίον αυτών των ανθρώπων. Μπορείτε να βασιστείτε στον Νταβίτ Κάσα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την αποστολή μας ε, στην Μάλτα. Υπάρχουν αρκετά ε, στοιχεία στην αναφορά. Στην έκθεση υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές κατηγορίες οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν. Η έκθεση και η σημερινή συζήτηση δείχνουν λοιπόν ότι πρέπει να γίνει ακόμα αρκετή δουλειά. Δείχνει ταυτόχρονα ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν αντικατοπτρίζει ε, μονάχα μία άποψη ε, και ε, οι άποψεις, άποψεις στην Μάλτα είναι πάρα πολύ πολλωμένες για να έχουμε μία συνολική εικόνα. Καθημερινά λαμβάνουμε καινούργιε πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Δυστυχώς όμως δεν είμαστε ερευνητές αστυνομικοί. Κάνουμε τις συστάσεις μας Όμω ε, θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητη και υπεύθυνη δουλειά των αρχών της ε, Μάλτας και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι ιδιαίτερω για το, το λόγο ε, ότι ο Υπουργό Δικαιοσύνη βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα και ότι έχει συναντήσει κάποιους από τους εκπροσώπους μαζί μας οι οποίοι δεν έχουν λάβει όλες τις απαντήσεις και εγώ έχω κάποια ερωτήματα, για, παραδείγματα, για παραδείγμα ποια μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση για να μπορέσει να ενισχύσει την ανεξαρτησία ε, της ε, δικαιοσύνης, ε, πώς το σύστημα των εισαγγελέων λειτουργεί στην Μάλτα εάν ασχολήθηκαν με, τις, με τα ζητήματα τα οποία αφορούσαν ε, την ε, κυρία Γκαλίτσια. Επίσης, μαζί μας είναι η γη της κυρίας ε, Γκαλίτσια. Πρόσφατα τους φιλοξένησα και σε μια εκδήλωση του Κοινοβουλίου όπου συζητήσαμε την ελευθερία του τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεισφορά τους ήταν πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε τα στοιχεία και θα συνεχίσουμε τον διάλογο με όλους όσοι ενδιαφέρονται για την κατάσταση στη Μάλτα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζάβιτς, παρακαλώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, ε χαιρετίζοντας ε, τον Άντρου ε, και τον Μάθιου, τους γιους της Δάφνης. Η δολοφονία της μητέρας σας δεν ήταν απλά μια δολοφονία για να σοπάσει έναν άνθρωπο ο οποίος πάντα με μεγάλο θάρρος προσπαθούσε να φέρει στο φως την αλήθεια. Ταυτόχρονα ήταν και μια επίθεση στην ελευθερία μας του, του λόγου και του τύπου διότι είναι μια ελευθερία η οποία διασφαλίζει ότι θα ακολουθήσουμε αυτό το οποίο προσπάθησε να ε, κάνει η Δάφνη. Ε, προσπάθησε να καταπολεμήσει περιπτώσεις διαφορές, τι τις οποίες συζητή, συζητούμε σήμερα εδώ. Ε, δεν μπορώ να μην αφήσω ασχολίαστη την αδιαφορία της, ε, δικαιούς, της κυβέρνησης, την αδράνεια της κυβέρνησης σε όλα όσα έχουν προκύψει από την Επιτροπή η οποία οποία ε, επισκέφθηκε την ε, Μάλτα. Η απάντηση από τον Πρωθυπουργό της Μάλτας ήταν ότι ε, φροντίζει μονάχα ότι λένε οι υπουργοί στη Μάλτα και όχι οι ευρωβουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αγνοεί τη φωνή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα βέλτιστα για να υπερασπιστούμε την ελευθερία του τύπου και επίσης παρουσιάσαμε και έναν ε, νόμο στην ε, ε, πρακτική αυτή όπου τράπεζες όπως οι πιλάτες θα μπορούν να σταματήσουν τη λειτουργία τους και οι δράσεις ε, που γίνονται κατά ε, τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα σταματήσουν. Είναι πολλές σοβαρές δράσεις τις οποίες θα πρέπει να ξεκινήσουμε διότι όταν σοπαίνουμε τον τύπο τότε κάνουμε επίθεση στους, πολίτες, στους Ευρωπαίους πολίτες κάτι το οποίο είναι σημαντικό για εμάς. Ευχαριστούμε συνάδελφοι για το ότι τηρήσατε το χρόνο και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Υπουργό. Να έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν που επίσης έχει κάποια ερωτήματα, έχει λάβει κάποια ερωτήματα, όμως ε, παρακαλείστε να είστε ε, σύντομοι και να απαντήσετε μέσα σε δύο λεπτά. Ε, Υπουργέ Μπονίτσι, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε την ευκαιρία να παρευρεθώ εδώ σήμερα και να συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί σα. Φυσικά, σε πέντε λεπτά δεν ε, δίναμε να απαντήσω όλε τι ερωτήσει σα, αλλά ούτε καν ένα τμήμα εξ αυτών, αλλά είμαι ανα πάσα στιγμή πρόθυμο να ξαναέλθω εδώ για να απαντήσω οτιδήποτε ερώτηση θέλετε να απαντήσω. ω κυβέρνηση, σκοπός μας είναι να δώσουμε τη σωστή εικόνα της Μάλτα την εικόνα την οποία συζητήσατε εδώ πέρα σήμερα δεν είναι πραγματική εικόνα της Μάλτας. Δεν είναι σωστή αυτή η εικόνα της Μάλτας και θέλουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το διάλογο για να δώσουμε τη σωστή εικόνα της χώρας. Για να σας δώσω λοιπόν ποια είναι η εικόνα, μια εντύπωση. Λίγες ημέρες μετά την ε, φρικτή δολοφονία της Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια που σόκαρε όλους ε, μας στη Μάλτα και σε όλη την Ευρώπη και φυσικά ε, θέλω να δώσω τα συλλαλπιτήριά μου στην οικογένεια της Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια. Κατανοώ την οργή τους, κατανοώ τα συναισθήματά τους σήμερα και τις τελευταίες ημέρες μας συγκλώνησε μα συγκλώνησε η δολοφονία αυτή. Μετά από λίγες ημέρε λοιπόν μετά την δολοφονία, μία από τι βασικές εφημερίδες έκανε μία έρευνα για το κράτο δικαίου και ρώτησαν τον κόσμο και μιλάμε για μια κυβέρνηση, μια εφημερίδα η οποία συνήθω είναι πολύ επικριτική για την κυβέρνηση, Sunday Times of Malta ονομάζεται. Ζήτησαν λοιπόν το, από τον κόσμο να πει κατά πόσον ε, εμπιστεύεται τι αναπλέ δυνάμει τη Μάλτα. 72% είπαν ναι, εμπιστεύεστε την κυβέρνηση. 72% είπαν ναι, εμπιστεύεστε την αστυνομία. 69% είπαν ότι ναι, εμπιστευόμαστε την αστυνομία. Εμπιστεύεστε τα μέσα ενημέρωση. 51% είπαν ναι. Αυτό είναι λοιπόν μια, ένα στιγμιότυπο τη έρευνα αυτή τη εφημερίδα και των αποτελεσμάτων. Να επανέλθω στην έκθεση λοιπόν που δυστυχώς ε, θεωρώ ότι δεν ε, κατανοεί το ρόλο των θεσμικών οργάνων στη Μάλτα που περιγράφει το πώς αυτά τα θεσμικά όργανα ε, εκτελούν τα καθήκοντά τους. Αυτό που είναι ακόμα χειρότερο είναι το εξής, ότι οι υπεύθυνοι για την σύσταση της έκθεσης αυτής χρησιμοποιούν συστάσεις οι οποίες είναι είτε παροχημένες χρονικά, είτε αναλυθεί σε ό,τι αφορά τα θεσμικά όργανα της Μάλτας για τις αποφάσεις που έλαβε η Μαλτέσικη κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι και άλλα κρατημέλη λειτουργούν με τα ίδιο σύστημα και έχουν λάβει παρόμοιες απαντήσεις. Αποφάσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Έχω ολόκληρο κατάλογο μεταρρυθμίσεων που έχουμε κάνει τα τελευταία πέντε χρόνια και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας αυτές με κάθε δέσμευση, με κάθε επιμέλεια. Αυτό δεν έχει τονιστεί επαρκώ ε, στην έκθεση τη αποστολή ένα από του συναδέλφου σα λοιπόν με ρώτησε το εξή. Ναι, ε, συγγνώμη, εγώ δεν σα διέκοψα. Ούτε βρίσκομαι εδώ να τσακωθούμε. Ε, ήρθα εδώ για να σα μιλήσω, να απαντήσω στα ερωτήματά σα ανά πάσα στιγμή όπου θέλετε. Είμαστε πρόθυμοι και ανοιχτοί για επικοδομητική συζήτηση. Είμαστε εδώ ως κυβέρνηση που θέλουμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να προωθήσουμε την πραγματική εικόνα της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος λοιπόν με ρώτησε, Υπουργέ, πείτε μας, οι αιτιάσεις, οι πιο σοβαρές αιτιάσεις ερευνώνται, ερευνώνται. Η απάντηση είναι ναι. Στη Μάλτα έχουμε ένα σύστημα που οποιοδήποτε μπορεί να φέρει πληροφορίες σε οποιοδήποτε δικαστήριο και το δικαστήριο μπορεί να ερευνήσει οποιαδήποτε πληροφορία του χορηγήσει ο οποιοδήποτε πολίτης. Όλα τα βασικά ζητήματα, όλες οι βασικές αιτιάσεις οι οποίες ε, κατέγγειλε η Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια βρίσκονται υπό έρευνα από το δικαστικό σώμα, συμπεριλαμβανομένης και μίας αιτίασης, πάρα πολύ σοβαρής, ε, την οποία ο, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος ζήτησε από το δικαστικό σώμα να ερευνήσει. Όταν λοιπόν έρχεστε και μου λέτε ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου και δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει διαφάνεια στη Μάλτα, πρέπει απλά να σα πω ότι αυτό δεν αληθεύει, δεν στέκει, γιατί όλε οι βασικές κατηγορίες είναι υπό έρευνα από το δικαστικό σώμα. Κατόπιν ε, αιτήματο είτε του πρώην ε, επικεφαλής της αντιπολίτευσης ή του Πρωθυπουργού. Τώρα, να σας μιλήσω για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Η ιδέα ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πετάξει στο σκουπίδι το κράτος δικαίου είναι πραγματικά άδικη και δεν στέκει. Η πολιτική λοιπόν στη Μάλτα. Αν κρυθούν ότι έχουν διαπράξει πράξεις διαφθοράς θα συνεχίσουν να διώκονται για όλη τους τη ζωή. Εφόρου ζωής. Πείτε μου, μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει τέτοια νομοθεσία. Επίσης έχουμε μία νομοθεσία για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Και λυπάμαι, πρέπει να σας πω ότι η κυρία Γκόμες, την οποία και σέβομαι, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει απόλυτα πώς λειτουργεί η νομοθεσία για τους πληροφοριοδότες. Δεν νομίζω ότι φταίει γι' αυτό, γιατί η προστασία των πληροφοριοδοτών ε, είναι σπάνιο ως νομοθεσία να υπάρχει στην Ευρώπη. Η Μάλτα θεωρώ και ενδεχομένω άντε άλλα δύο-τρία κράτη να έχουν τέτοια νομοθεσία. Προκειμένου λοιπόν ένα άτομο να έχει το καθεστώ προστασία, θα πρέπει να προβεί σε κάποια αποκάλυψη. Αυτό είναι εγγενέ. Έτσι λειτουργεί ο μηχανισμό προστασίας των πληροφοριοδότων. Όταν προβεί λοιπόν σε κάποια αποκάλυψη, αυτόματα λαμβάνει προστασία. Στην περίπτωση λοιπόν του κύριου Φέρε, ο οποίο πρέπει να σας πω ότι η κυρία Εφεμόβα, η οποία επίσης αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, είχε πολλές ε, επιφυλάξεις γι' αυτόν. Ο κύριος Φέρε λοιπόν θέλει να έχει προστασία ω πληροφοριοδότη, γιατί σκοπεύει να ζητήσει άμα ασυλία από την εισαγγελία. για πληροφορίες που απαγορεύεται από το FIU να δημοσιευτούν. Υπάρχει αυτή η αρχή η οποία διέπει όλες τις αρχές ε, σε ό,τι αφορά τις ε, χρηματοοικονομικές εισαλλαγές που απαγορεύει τη δημοσίευση απορτών πληροφοριών. Ο κ. Φέρης θέλει να καταγγείλει, θέλει να παραβιάσει αυτή τη ρήτρα και θέλει να χρησιμοποιήσει την προστασία του ως πληροφοριοδότη. Έχω κι άλλα να αναφέρω πολλά, αλλά ναι, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας ε, ζητήσω να ολοκληρώνετε. Αλλά πολύ απλά δεν δέχομαι αυτή την ε, λαθασμένη εικόνα που δόθηκε γιατί η Μάλτα δεν προσπαθεί να προωθήσει το κράτος δικαίου. Καταρχάς, να σας πω κάτι άλλο δημιουργήσαμε μια επιτροπή. Εμείς δημιουργήσαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή που περιλαμβάνει και τον επικεφαλής του δικαστικού σώματος που δίνει συστάσεις για τις, ε, τους διορισμούς στο δικαστικό σώμα. Αυτή ήταν δική μας μεταρρύθμιση. Επίσης, ε, περάσαμε την ε, τέταρτη οδηγία κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Δεν ισχύει ότι δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η τέταρτη οδηγία στην ε, νομοθεσία μας. Το συντομότερο δυνατόν μετά τις εκλογές, γιατί έγιναν εκλογές τον Ιούνιο. Και αυτό πλέον περιλαμβάνεται, είναι τμήμα του συντάγματός μας. Κάτι άλλο που ήθελα να υποδείξω. Ε, υπήρξαν διάφορες ε, αιτιάσεις εδώ ότι η Μάλτα αντιμετωπίζει ε, Στη Μάλτα υπάρχουν υπόνοιες, σαφείς υπόνοιες ακούστηκαν ότι η Μάλτα ε, υποσκάπτει το κράτος δικαίου και δεν σέβεται τις ευρωπαϊκές αρχές. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ομοφωνία και από τον ε, Πρωθυπουργό και του επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Μάλτα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Χθε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Μάλτα είπε με σαφήνεια ότι είναι κατά της ε, υπόνοια αυτή ότι υπάρχει βασικός κίνδυνος, σημαντικός κίνδυνος παραβίασης του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών, αρχι... των ευρωπαϊκών αρχών, σε ό,τι αφορά και το άρθρο 7 ε, στη Μάλτα. Αυτά ήθελα να πω λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ζητήσω από τους ευρωβουλευτές να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Είμαστε εδώ για να σας δώσουμε την πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει στη Μάλτα και το τι κάνουμε για να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου, το οποίο είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και αποτελεί τη βάση της δημοκρατίας τη βάση των ευρωπαϊκών αρχών και είναι και ο λόγος άλλωστε που και εγώ και η υπόλοιπη κυβέρνηση αφιερώνουμε τις καριέρες μας για να βελτιώσουμε και να κάνουμε καλύτερο μέρος στην Ευρώπη. Ο κύριος Γκίγκολτ, θα ήθελα να σας πούμε ότι θεωρούμε ότι όλες αυτές οι δηλώσεις είναι αναλυθείς και δεν στέκουν. Σας παρακαλώ, ζητώ τάξη, λέει η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Γκάλα. Ο κύριος ε, Αριστοτέλης Καρτσιάδης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δύο λεπτά παρακαλώ για να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Ε, first... Ε, Όσον αφορά την οδηγία καταπολέμησης νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων, μετεφέρθη το Δεκέμβριο του 2017. Επομένως, η εφαρμογή είναι τελείως διαφορετική υπόθεση, η μεταφορά είναι κάτι άλλο. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας. Όσον αφορά τις δύο ερωτήσεις της κυρίας Σίνεντβελτ, η πρώτη όσον αφορά την υπηκότητα μέσω επενδυτικών προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά αυτά τα επενδυτικά προγράμματα και το πώς δίνεται η θαγένεια ε, σε όλες τις χώρες, ε, συμπεριλαμβανομένες και της Μάλτας. Ε, σε όλα τα θέματα ε, στα οποία θα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις για να δοθεί η υπηκότητα, θα πρέπει να υπάρχει στενή σχέση ε, μεταξύ της αίτησης και του ετούντος και της χώρας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Μάλτα κατέληξε σε συμφωνία τον Ιανουάριο του 2014 για το πρόγραμμά της και υπήρχε υποχρέωση να δείχνουν ότι υπάρχει κατοικία και αυθεντική σχέση με τη Μάλτα πριν τους δοθεί η υπηκότητα. Όσον αφορά το θέμα της διαφθοράς, πράγματι η ετήσια έκθεση διαφθοράς δεν υπάρχει πλέον, αλλά επίσης για πρώτη φορά φέτος, και αυτό σας το διαβεβαιώ, θα υπάρξει ένα πολύ εκτεταμένο τμήμα που αφορά τη διαφθορά στην ε, ετήσια έκθεση για τη Μάλτα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, γιους της Δάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια. Καλώς ορίσατε εδώ στην Επιτροπή μας. Έχετε δύο λεπτά για να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή που μας δίνετε το λόγο. Δεν περιμέναμε να μιλήσουμε. Ο αδερφός μου και εγώ ήρθαμε εδώ σήμερα απλώς για να δείξουμε την υποστήριξή μας. Διεκδικήσουμε τα βασικά μας δικαιώματα. Ε, υπάρχει υπόθεση ενώπιον του Μαλτέζικου Δικαστηρίου για να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα την οποία ε, προσπαθεί να παρακολύσει η κυβέρνηση. Αλλά για μας ε, το θέμα δεν είναι μόνο η έρευνα για τη δολοφονία της μητέρα μας. Αυτό είναι αυτό το οποίο πήγε περισσότερο γιατί ο φόβος μας καθημερινά εξαφανίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία ο άνθρωπος αρμόδιος ε, για την ε, αστυνομική για έρευνα είναι κάποιος τον οποίο ερευνούσε η μητέρα μου. Ο δικαστής είναι κάποιος που ερευνούσε η μητέρα μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να εμπιστευτούμε τους θεσμούς της χώρας μας όταν οι άνθρωποι που ερευνούσε η μητέρα μου για πάρα πολύ σοβαρά δικήματα εξακολουθούν να προσπάθησε να κάνει η μητέρα μας να μην εξαφανιστεί και να μην ξεχαστεί. Και τα όσα κάνατε εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο ε, ελαφραίνει λίγο το βάρος στους ώμους μας. Ε, για παράδειγμα, σε άσπρο μαύρο ε, στην έκθεσή σας. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς ε, πλέον. Η μητέρα μας έχει πεθάνει, αλλά τουλάχιστον μέσω του έργου σας ζει και αν σταματήσετε τη δουλειά σα, εμεί δεν θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε, αλλά θα είναι πολύ πιο δύσκολο για μα. Το μήνυμά μα λοιπόν προ εσά είναι μην αφήσετε πιο ε, φιλικά προσκύμενο. Ο αδερφός μου και εγώ δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε καμία σχέση με την κυβέρνηση, τουλάχιστον ε, με τα κόμματα που βρίσκονται στην ηγεσία. Εμά και είναι μια ε, χώρα που έχει γίνει η πίσω πόρτα τη Σέγγεν. κανει δεν αγοράζει, δεν ελέγχει ποιο αγοράζει διαβατήρια. Για παράδειγμα, πώ ένα Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαστε μεν εμπειρογνώμονε ε, στα όσα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είμαστε βέβαιοι τι εργαλεία έχετε στη διάθεσή σα. Δεν είστε ανακριτέ ερευνητέ, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά πιέζετε και όσο περισσότερο πιέζετε, τόσο υπόλογη θα είναι η κυβέρνησή μα, τόσο πιο υπόλογη θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν σας προτρέπουμε να μην αποφασίσετε. Έχετε όλοι γίνει πλέον οι δήμονες στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μάλτα. Θα πω όμως ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται δικαστική. Τα στοιχεία αυτά μόνο όταν δόθηκαν στην αστυνομία, όταν η αστυνομία δεν έδρασε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επισημάνουμε σε ένα πλαίσιο όπου η ε, πληροφορία δεν τύχουμε. Thank you. Our thoughts and prayers are with you. Σας ευχαριστώ της προθυμίας του Υπουργού Μπονίτσι να απαντήσει και σε περαιτέρω ερωτήσεις που θα χρειαστεί ενδεχομένως. Ασφαλώς ζητήσαμε επίσης ε, με μέλη του δικαστικού σώματος να έρθουν στις Βρυξέλλες. Ζητήσαμε τεκμηρίωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι λομπίστες, έχουν ε, μέλη του λόμπι στις Βρυξέλλες. Τους καλέσαμε και αυτούς. Το μοναδικό για την αποστολή στις 31 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου. Και χαίρομαι πλέον ε, σε 15 λεπτά από το επόμενο θέμα τη σημερινή διάταξη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σα και την κατανόηση που δείχνετε. Και να ζητήσω από τον προσκεκλημένο μα, τον κύριο Γκόουσταϊλ και την κυρία Λάγκμπακ, να έλθουν εδώ. <laughs> Σας παρακαλώ, οι συζητήσεις εκτός αιθούσης. So, uh, εξάρτηση και την κυρία Βιτσίνσαν Ντέντλε, η οποία είναι υπεύθυνη για θέματα ισότητας. Όπως ξέρετε, εργαζόμαστε στον τομέα. Έχουμε ένα δίκτυο για την ε, βελτίωση της συνεργασίας ε, στο, στο ΜΙΣ ε, κοινού ενδιαφέροντος. Η ετήσια έκταση του 2017 για τη συνεργασία του δικτύου το 2017, ο κ. Γκούστελ θα μας παρουσιάσει τις βασικά επιτεύγματα του 2017. Θα δώσουμε το λόγο στη συνέχεια στην κυρία Λάγκμπακ για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της συνεργασίας, όπως συμφωνήθηκαν για, τα, για τις υπηρεσίες το 2018. Και μια και είναι μαζί μα η κυρία Λάγκμπακ σήμερα, πλήσατε από την Επιτροπή ΦΕΜ. Να δώσω το λόγο καταρχά στον κύριο Γκούστελ. Θα μπορούσατε να είσαστε σύντομο, γιατί έχουμε χάσει χρόνο στο προηγούμενο θέμα. Επτά λεπτά έχετε στη διάθεσή Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, καλημέρα κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι ε, τιμή ε, το γεγονός ότι μπορώ να σας παρουσιάσω σήμερα τα αποτελέσματα ε, της έκθεσης του Δικτύου Ευρωπαϊκών Οργανισμών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης. Ήμουνα πρόεδρος του Δικτύου πέρυσι για το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Το δίκτυο υπάρχει λόγω της ανάγκης ε, για πραγματική συνεργασία και γι' αυτό το λόγο ε, υπάρχει το συγκεκριμένο ε, όργανο. Ήμασταν ιδιαίτερα ενεργοί και ο ρόλος της Προεδρίας του Δικτύου είναι να συμβάλλει στη συνεργασία καθώς επίσης και να προτείνει διάφορα κοινά προγράμματα, μερικά εκ των οποίων θα σας παρουσιαστούν εν ολίγες. Ε, αρχικά θα ήθελα να σας ε, μεταφέρω ένα μήνυμα ε, των διευθυντών των Οργανισμών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή ε, εξετάζει πάντοτε ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ε, πόρων ε, και των αυξανόμενων προσδοκιών για, τις, για τους συγκεκριμένους οργανισμούς και όλο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη από εμάς κατά την προετοιμασία του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο θα είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit ε, και θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στον τομέα εσωτερικών υποθέσεων ε, και δικαιοσύνης. Ε, το δεύτερο το, για το οποίο θα ήθελα να σας ενημεράσω είναι ότι μία από τις βασικές προκλήσεις για τις υπηρεσίες είναι να ενισχύσουμε την ε, ε, διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων ε, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των εντολών που έχει ο κάθε οργανισμός και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη μας τη νέα νομοθεσία σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Παρ' όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα ε, έχουμε αρκετό έργο μπροστά μας ε, ε, και υπήρξαν αρκετές τεχνικές, τεχνικά επιτάευματα πέρσι. Το τρίτο θέμα αφορά ε, το γεγονό ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέε προκλήσεις, ε, την μετανάστευση αλλά και την ασφάλεια και τους ε, δεσμούς που έχουν με τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλέ, απαιτείται συνεργασία με τρίτε χώρε σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ποτέ πριν και οι υπηρεσίες έχουν οργανώσει μια πρώτη συνάντηση των υπευθύνων για τον συντανισμό και να εντοπίσουν του τομεί όπου θα μπορούσε να υπάρχει δυνατότητα στενότερης ε, συνεργασίας και συνεισφοράς από τις υπηρεσίες μας. Αυτό είναι τα ε, τρία ε, βασικά μηνύματα και τώρα κάποιες πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά μηνύματα και τώρα ε, κάποιες πιο πρόσφατες ε, πληροφορίες ε, σχετικά με, τις, με ζητήματα συνεργασίας των οργανισμών όπως είναι για παράδειγμα η χρήση του κυβερνοχώρου για εγκληματικές παράδειγμα το γεγονός ότι ακόμα θα πρέπει να προσαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο στην ψηφιακή εποχή για παράδειγμα λοιπόν όταν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προσπαθούν να καταπολεμήσουν το κυβερνοέγκλημα, το οποίο είναι υπερεθνικό εκφύσεως. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταυτοποιήσουμε ε, και αν, παρόλο που έχουν υπάρξει κάποιες βελτιώσεις και βήματα προς τα εμπρός, οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί είναι ακόμα διατεθειμένοι να παράσχουν τις βοήθεια για να καλυφθούν αυτά τα προβλήματα. Ε, λέγοντας αυτά είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται δικαιοσύνη και οι ε, αστυνομικές αρχές θα πρέπει να έχουν τα αναγκαία εργαλεία. Έχουν υπάρξει σημαντικές έρευνες στα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια ε, και θα πρέπει να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Η σημασία ενίσχυσης ε, της ε, συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι το, το πλαίσιο θα υπάρξει μια τεχνική συνάντηση με την βιομηχανία και τους οργανισμούς το ε, θέμα ε, του ε, εκπαίδευσης σε διάφορους τομείς και νέα ειδίκευσης έχει συζητηθεί διότι προσφέρονται μόνο και σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις και και όχι μονάχα όσον αφορά εργαλεία και μεθοδολογία αλλά και την πρόσβαση στα εργαλεία τα οποία χρειάζονται για να γίνεται η δουλειά Εξέχασα τώρα την, το γεγονός, η νέα αναφορά, η νέα έκθεση την οποία παρουσιάσαμε πέρσι ήταν μια κοινή έρευνα σχετικά με το σκοτεινό ε, δίκτυο, με το Darknet, ε, όπου υπάρχει μια ε, λεπτομερής ανάλυση σχετικά με τα πιο, με τις, με με πιο είχαμε αρκετές ε, πρωτοβουλίες. Ε, η Frontex ε, ανέλαβε την πρωτοβουλία για να δημιουργήσει δύο ζητήματα, δύο κινήσεις ε, για την ε, μετανάστευση. Ένα νέο ε, θέμα το οποίο εισήχθη από το Κέντρο Παραγωγικών Μεταναστών ενώ επίσης η εκπαίδευση του προσωπικού ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης είναι κάτι το οποίο το κάνουμε όλοι εμείς και ο δικός μας ο οργανισμός ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα των μεταναστών. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν όμως κάποια θέματα τα οποία Ένα από τα θέματα τα οποία προεκύψαν από συζητήσει με τους οργανισμούς είναι το γεγονός ότι ε, το ζήτημα της υγείας ε, θα πρέπει ε, να συνεχιστεί και στο, να δοθεί και στο προσωπικό το οποίο εργάζεται για τους οργανισμούς. Και τώρα το τελευταίο σημείο, το οποίο εργασία και την ε, πρόληψη. Έχουμε εντοπίσει ε, ασθένειε, ζητήματα ασθενειών ε, και η έρευνα που πρέπει να γίνεται, καθώς επίσης και κατευθυντήριε, οι οποίε δεν είναι πάντοτε διαθέσιμε ε, στα, hot, spots και γι' αυτό το λόγο δίνεται εκπαίδευση, παράσχεται εκπαίδευση στο προσωπικό για να μπορέσει με τι παρεμβάσει. μπορείτε να το δείτε στη διαφάνεια. Και εδώ μια τελευταία φωτογραφία με την ομάδα των διευθυντών ε, και επίσης είχαμε ε, τον ε, Γενικό Διευθυντή Δικαιοσύνης εδώ πέρα και ε, το μήνυμα που μπορώ να σας μεταφέρω λοιπόν ε, και ε, η συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο έχει δείξει ότι το δίκτυο έχει οριμάσει και επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα έργα τα οποία θα πρέπει να εκπληρώσουν με βάση την εντολή τους οι οργανισμοί και να βοηθήσει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, θα χαρώ να ε, παραδώσω τώρα τα κλειδιά της ευθύνες στον κύριο Λάγκμπαχ, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων και θα έχει την ενέργεια για να προωθήσει όλα αυτά και να λαμβάνει υπόψη του ζητήματα τα οποία είναι μεταξύ άλλων η ευθύνη των οργανισμών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούσπτα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και σας ευχαριστώ και για τη δουλειά που κάνατε ως ε, επικεφαλή σε αυτό το δίκτυο στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λάγκπακ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Προσπαθήστε και εσείς να τηρήσετε το ε, Θα ήθελα να σας ζητήσω να σκεφτείτε την τελευταία φωτογραφία που σας έδειξε ο Αλέξης, ε, όσον αφορά την ε, ισότητα των φύλων, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη συνεδρίαση και όταν ε, βλέπετε ότι από τους εννέα διευθυντές υπηρεσιών αυτή τη στιγμή είμαι η μόνη γυναίκα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο χρειάζεται και η δουλειά μας, ίσως να συζητηθεί και το θέμα αυτό και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Σύντομα θα είμαστε δύο γυναίκες διευθύντριες. Ε, θα σας πω λίγα περισσότερα εντός ολίγου για τα νέα πράγματα τα οποία θα φέρουμε εμείς ε, στο έργο της ε, κοινή σύμπραξης αυτών των εννέα υπηρεσιών. Αλλά όπως γνωρίζετε, εμείς είμαστε η μόνη υπηρεσία μεταξύ των εννέα που δεν είναι υπό τη, σκέψη της, υπό τη της ΛΥΜΠΕ. Είμαστε υπό τη σκέπη της Επιτροπής Γυναικών. Το γεγονός λοιπόν ότι θα προεδρεύουμε εμείς του δικτύου έχει και νέες συνέργειες. Θα γίνονται συνεδριάσεις φυσικά με την Επιτροπή Γυναικών. Αλλά κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας του των ε, ε, υπηρεσιών ε, θα είναι και Επιτροπή Γυναικών Αρμόδια. Ο Αλέξης μας είπε τι κάνουν οι υπηρεσίες και το βασικό μήνυμα είναι ότι εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία. Όχι μόνον για το Κοινοβούλιο, όχι μόνον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κυρίως για τους χρήστες. Και όπως γνωρίζετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες και το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές ε, επικεντρώνονται στην ασφάλεια και στη δικαιοσύνη και η πλειοψηφία των υπηρεσιών είναι αυτές οι οποίες ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Εμείς κυρίως επικεντρώνουμε ε, τις προσπάθειές μας στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των έσω. Ε, βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τόσο πολύ τους άλλους οργανισμούς για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, αλλά καταρχάς θα συνεχίσουμε τη δουλειά που ήδη ξεκίνησε και την ανέφερε και ο Αλέξης προηγουμένως ε, την προηγούμενη χρονιά, και επειδή εμείς είμαστε πάρα πολύ μικρή υπηρεσία, είμαστε πιο μικροί από όλου ε, και συμφώνησαν και άλλοι συνάδελφοι ότι η ΣΕΠΟΛ, η Αστυνομική Ακαδημία, θα συνεχίσει να συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Και εμείς ε, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα προσθέσουμε περισσότερα για τη βία κατά των γυναικών και τη την ε, οπτική των στατιστικών βάση φύλου. Αυτή είναι η δική μας νέα συμβολή. Και επίσης ε, η Frontex θα συνεχίσει να είναι επικεφαλής για όλα τα θέματα που αφορούν τη μετανάστευση, τη διαχείριση συνόρων κλπ. Όλα αυτά τα θέματα δεν έχουν επιληθεί ακόμα, χρήζουν ακόμα δουλειά και είναι πολύ σημαντικό αυτή Η λειτουργικότητα των ε, συστημάτων πληροφορικής, κάτι που αναφέρθηκε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτό που θα συζητήσουμε τώρα όμως είναι τι θα συμβάλλουμε εμείς. Νομίζω ότι για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσει καταρχάς ε, αυτό το ποιες υπάρχουν και πώς, διαφορετικά, πώς επιδρούν αυτά διαφορετικά σε αυτούς. Πώς μπορούν να διαφοροποιήσουν τα πράγματα οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, για να Υπάρχει αποτελεσματικό σχεδιασμό των μέτρων. Ε, υπάρχει αντίκτυπο σε όλου του τομεί. Κοιτάμε να δούμε λοιπόν πώ θα είναι αυτό ο αντίκτυπο. Τι είναι τα στατιστικά φύλου. Είναι τελείω διαφορετικά. Στατιστικά καταμερισμένα αναφύλλω και από εκεί και πέρα έχουμε στατιστικά ε, φύλου gender statistics. Επομένως, και θα εκπαιδευτούμε, θα επιμορφωθούμε, αλλά θα έχουμε και μία προσέγγιση για να δούμε πώς ε, έγινε η επιλογή. Θα σας δείξουμε μέχρι το τέλος του έτους πώς ε, ενώ, ε, τομέα θα έχουμε την ψηφιοποίηση, διότι ε, τουλάχιστον από πλευρά φίλου δεν είναι μόνο προτεραιότητα της ε, Βουλγαρικής, αλλά και η Αυστριακή Προεδρία στη συνέχεια θέλουν να ασχοληθούν με την ψηφιοποίηση και τις τεχνολογίες από τη σκοπιά του φίλου. Και αυτό φυσικά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε πώς ε, και οικογενειακού βίου. Θα σας επιτρέψουμε έτσι να λάβετε μια μικρή ματιά. Και ξέρω ότι ίσω δεν είχατε χρόνο, αλλά θα ήθελα να πω με ιδιαίτερη περηφάνεια ότι όλοι οι διευθυντέ υπηρεσιών και ο Αλέξη ε, και όλοι οι υπόλοιποι διευθυντέ υπηρεσιών στη Λισαβόνα όταν συναντήθηκαν συμφώνησαν. Okay. Τα αγγλικά θα βρίσκεται στο 2, στο κανάλι Παριθμό 2. Μάλιστα. Για τρίτη φορά λοιπόν και ελπίζω τώρα να με ακούτε. Χαίρομαι λοιπόν που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα αυτή, η ανταλλαγή πληροφοριών μάλλον και χαίρομαι που έχουμε ε, ισότητα φίλων εδώ. Έχουμε ίσο ρυθμό γυναικών και ανδρών. Μας αναφέρατε τα θέματα που σας απασχολούν στις εργασίες σας. Να αναφερθώ σε αυτό που είπατε για τα νέα εργαλεία για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Είπατε ότι θα πρέπει να βρούμε νέα εργαλεία για να εντοπίζουμε τα κυβερνοεγκλήματα. Μίλησατε για συμπράξεις δημοσίου και δυτικού τομέα. Δεν πιστεύω όμως ότι αυτά, παρόλο που είναι σωστά και καλά, αρκούν. Έχετε περαιτέρω μέτρα κατά νου, περαιτέρω εργαλεία για τον εντοπισμό κυβερνοεγκλημάτων. Μιλήσατε επίσης για την υγεία στον χώρο εργασίας και τα γενικά αυτά πρότυπα. Έχουμε παντού τα απαραίτητα εργαλεία για να ερευνούμε τα φαινόμενα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό να μην υπάρχουν μόνο κανόνε, αλλά να υπάρχει και σωστό εξοπλισμό σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Ασφαλώ συμφωνώ μαζί σα. Και ακόμα πριν το πείτε, είχα προσέξει ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερη ισότητα φύλων στη φωτογραφία αυτή. Αυτό προφανώ. Το θέμα της η ισότητα των φίλων πάντα αποτελεί αντικείμενο προστιθέμενης αξίας, γιατί και από τροπολογικής άποψης οι γυναίκες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εγγενώς, τα οποία μπορούν να ωφελήσουν κάθε κλάδο Θα πρέπει λοιπόν να στραφούμε προς την ισότητα των φύλων για να πετύχουμε πιο πολύ αξία. Ελπίζουμε λοιπόν να έχετε πάνω από δύο γυναίκες ε, στην ομάδα σας και ελπίζουμε να συνεργαστείτε και με την Επιτροπή Λίπε, γιατί Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσουμε και τους ε, πολίτες στην πατρίδα μας για τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. όλων των υπηρεσιών επί της σωστής βάσης είναι σαφές τώρα και είναι σαφές και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες για το μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία παρουσιάσατε είναι σημαντικά. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο στην ΛΥΜΠΕ για την παρουσίαση των πολυτομιακών δραστηριοτήτων και μέτρων με συνεπτικό τρόπο. Τρία σχόλια θα ήθελα να κάνω και για το MCDDA για τους τομείς που εμπλέκονται σε ό,τι αφορά τη συνεργασία. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη χρήση νέοπληση της, ε, των κυκλωμάτων ναρκωτικών είναι σαφέ ότι είναι απαραίτητο αυτό, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε το φαινόμενο για να το καταπολεμήσουμε. Ένα άλλο θέμα, ένα δεύτερο θέμα, έχει να κάνει με το ζήτημα των ναρκωτικών μεταξύ προσφύγων. Για να κλείσουμε τα σύνορα, πρέπει απλά οι πολιτικές μας να προσαρμοστούν στους πρόσφυγες. Αλλά από την άλλη είναι σημαντικό να υπάρχει και μια τέτοια ανάλυση, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την υγεία των ανθρώπων αυτών. Ένα τρίτο σημείο έχει να κάνει με την προετοιμασία, να κάνει και με το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης για τις νέες ψυχοτρόπες ουσία. Αν θα μπορούσατε να μας περιγράψετε εν συντομία το πώς προχωράνε οι προετοιμασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Χέιντε. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Ασχολήθηκα λίγο με το θέμα αυτό και νομίζω ότι μπορώ να σας πω κάποια πράγματα όσον αφορά την ισότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπε και ο συνάδελφος, δεν μπορούμε απλώς να μιλάμε για την ισότητα φίλων στην Επιτροπή των Γυναικών. Πρέπει να υπάρχει ισότητα σε όλες τις Επιτροπές. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να πω ότι ε, εδώ και 14 χρόνια εγώ δίνω μάχη για να ενταχθούν αυτά τα θέματα του φίλου σε όλες τις επιτροπές όχι μόνο επειδή υπάρχουν ε, δεσμευτικές εκθέσεις, αλλά για να υπάρχει πάντα η προοπτική του φέιλου και λειτουργήσε. Η ισότητα είναι κάτι το οποίο ε, προσπαθήσαμε να εντάξουμε και σπήραμε και πλέον έχουμε αρχίσει να απολαμβάνουμε τους καρπούς. Και ε, θα ήθελα και εγώ, όπως και ο συνάδελφος Μπόνι, ε, να πω το εξή. Ναι, έχουμε όλο ένα και περισσότερες γυναίκες σε ψηλά ιστάμενες θέσεις, αλλά δεν είναι πάντα τα πράγματα τόσο εύκολα. Ε, θα μας άρεσε να υπάρχει ισότητα παντού, αλλά είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επαγρυπνούμε, να υπάρχει η πίεση και οι γυναίκες να μπορούν μπορούν να αναλάβουν σημαντικέ θέσεις. Τώρα, όσον αφορά τι ποσοστώσει, νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Όπως ε, σα είπα, η ερώτησή μου είναι η εξή. Το θέμα των στατιστικών στοιχείων του φίλου. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει τα στατιστικά στοιχεία αυτά ε, να τα δούμε και υπό το πρίσμα αυτών που πλήττονται από την όλη κατάσταση. Αν όντω συμβαίνει αυτό, είναι εξαιρετικό. Η κυρία αρχικά όσον αφορά την ε, καταπολέμηση της ε, παρενόχλησης ε, και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ε, έχουμε συζητήσεις με όλους τους οργανισμούς ε, της ε, Ένωσης διότι έτσι θα μπορέσουμε καλύτερα να εργαστούμε. Εμείς ως οργανισμοί ακολουθούμε το πλαίσιο ε, τους ε, κανονισμούς. Ε, σκοπεύουμε όμως να εργαστούμε πιο συγκεκριμένα στην πιο απλή φύση όπως είναι για παράδειγμα σύμβουλοι που υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες. Όμως εμείς καθότι είμαστε ένας οργανισμός για την ισότητα των φύλων είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι για αυτό το θέμα οπότε έχουμε πιο συγκεκριμένες καταρτήσεις για τους συμβούλους όλους μας ε, σχετικά ε, με την ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμβούλων. Θα γίνουν συζητήσεις επίσης σχετικά με το πώς το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να εργαστεί. Ετοιμάζουμε εσωτερικά έγγραφα σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τις προκαταλήψεις αυτές οι επιρροές που δεν τις κάνεις επίτηδες αλλά επηρεάζονται από στερεότυπα όπως ε, όλα αυτά λοιπόν ε, θα συζητηθούν δεν πρόκειται να δημιουργήσουμε, είμαστε σε καλό δρόμο. Ε, στην έκθεση επίση θα δείτε μια πιο αναλυτική λίστα δραστηριοτήτων, ε, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειε τώρα. Τώρα όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Μπόνι, το δεύτερο ερώτημα αφορούσε τα ναρκωτικά και οι ε, πρόσφυγε και οι μετανάστες συμμετείχαν πάνω από 45, περίπου 50 χώρες για θεματικές συζητήσεις σχετικά με τη μετανάστευση υπήρχε, υπάρχουν... Ξεκινάνε οι ψηφοφορίε. Καλημέρα συνάδελφοι. Να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Έχουμε ένα θέμα το οποίο θα προχωρήσουμε βάσει της απλοποιημένης διαδικασίας. Οι συντονιστές της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ απόφασαν στη συνεδρίασή τους στις 11 Ιανουαρίου ότι το θέμα αυτό, δηλαδή η αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων για την ταξινόμηση οχημάτων στην ε, ε, Πορτογαλία, η οποία βασίζεται στη λεγόμενη απόφαση Προύμ. Το Κοινοβούλιο είναι διατεθειμένο να ξεκινήσει μια ε, εκτελεστική απόφαση για την έναρξη της αυτομετωπιωμένης ανταλλαγή δεδομένων για την ταξινόμηση οχημάτων στην Πορτογαλία και αυτό θα γίνει με την απλοποιημένη διαδικασία. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Κοράο, ο οποίος ε, είναι αρμόδιο ηγητή για το θέμα. Παρακαλώ μια σύντομη παρέμβαση κύριε Κοράο. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Με την απόφαση αυτή το Συμβούλιο συνεχίζει τη λεγόμενη απόφαση ΠΡΟΥΜ για την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Εδώ θέλουμε να επιτρέψουμε στην Πορτογαλία να λαμβάνει και να δίνει προσωπικά δεδομένα μέσω αυτόματης οδού για την ταξινόμηση των οχημάτων. Από όσα προκύπτει από την ανάλυση, η Πορτογαλία έχει μεταφέρει σωστά στην εθνική της νομοθεσία τις γενικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Ε, στο ε, κεφάλαιο 6 έχουμε και τη λεγόμενη απόφαση ΠΡΟΥΜ. Ε, πέρσι ε, το Κοινοβούλιο έλαβε ε, έτοιμα διαβούλευσης εντών τριών μηνών και για να μπορέσουν να απαντήσουν εγκαίρως, οι συντονιστές αποφάσισαν να εργαστούν αποκλειστικά στα αγγλικά μέσω της απλοποιημένης διαδικασίας βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού για να ψηφίσουμε στην επόμενη σύνοδο του Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια. Εδώ προτείνω το Κοινοβούλιο να δώσει τη συγκατάθεσή του και να υποστηρίξει απαραίτητο ε, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αυτοματοποιημένη Ανταλλαγή Δεδομένων που δημιουργείται βάσει τη απόφαση ΠΡΟΥΜ. Ευχαριστώ πολύ. Η απόφαση να εγκριθεί χωρί τροπολογίε. Υπάρχει κάποιο ο οποίο έχει αντίρρηση. Αν όχι, ε, εγκρίνεται η προτινόμενη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πηγαίνουμε στην ψηφοφορία για το κεντρικό σύστημα για την ε, ε, ταυτοποίηση το σύστημα έκρηση. Πρόκειται για το σύστημα λοιπόν έκρηση της ΙΕΝ. Να ρωτήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ντάλτον, αν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ντάλτον. Πολύ σύντομα, κυρία Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι όλοι θέλουν να ψηφίσουν. Να ευχαριστήσω όλου του και συζητητέ για τη συνεργασία στο θέμα αυτό. Νομίζω όλε οι ομάδε ε, ε, μετακινήθηκαν λίγο από τι αρχικέ του ε, θέσει και νομίζω ότι πλέον έχουμε μια καλή δέσμη συμβαστικών προτάσεων. Ευχαριστώ όλου λοιπόν και προσβλέπω στην ψηφοφορία. Ευχαριστούμε κύριε Ντάλτον. Να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία λοιπόν. 47. Έρχεται η ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, είναι πιο εύκολο. Πέραση της ψηφοφορίας. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 117. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Λειτουργεί. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σύστημα. 118. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. απορρίπτεται. 119, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 127. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, παρακαλώ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 136. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 137. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 138. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 139. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 140. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 141, 142 και 143 είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 144 και 145 είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 153, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 155, άρχεται η ψηφοφορία. της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Συγγνώμη. Κοίταζα την επόμενη τροπολογία. Τροπολογία 166. Άρχεται η ψηφοφορία. ταυτόσιμε με την 167. Έχετε δίκιο. Επομένω ψηφίζουμε και τι δύο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία έχουμε ένα επιπλέον μέλο από το ΕΛΚ. Κάποιο από το ΕΛΚ θα πρέπει ε, να βγάλει την κάρτα του. Ξαναψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ τις 166-167. και Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκατόν άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 172. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και περνάμε στην τροπολογία. 178. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 4. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 185. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρεύθηκε. 186. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 187. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 188 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 193. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 194. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 199 και 200. Ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 201. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 202 και 203. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνονται. η 204 και 205. Ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. Οι 206 και 207. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 208 και 209. Ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 210. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 211. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. 212. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 213. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 214. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6β. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 234. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 235. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 236. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 237. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται η ισοψηφία. 238. Είναι γλωσσική, δεν την ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τη 239. Παρακαλώ ψηφίζετε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 240. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 241. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 243 τώρα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 30. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 244. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. 245. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 246. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. 247. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. Περνάμε στην 254. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. Και τώρα περνάμε στην 38. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 262. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 263 και 264. Ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 265. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 39. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 266. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 267. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 268. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 269. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. 270. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 271. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 272 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 273 ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. Τροπολογία 274 και η τροπολογία 40 που είναι ταυτόσιμες. Από κοινού λοιπόν τις ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 200, μάλλον συμβαστική 7 τώρα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 282. Ψηφίζουμε. Πέρας. Έγκρινεται. 283. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 284. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 43. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 285. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 286. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 288 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 289 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 291 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 290 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στις 2.92 ε, και 2.93, είναι ταυτόσιμες, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στις 44, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2.94. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.95. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.96. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.97. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.98. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 300. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 301. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 302. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 303. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται ε, 2 γνωμοδότησε πέρας εγκρίνεται και τώρα πάμε στην τροπολογία 306 άρχεται πέρας απορρίπτεται συμβιβαστική νέα άρχεται πέρας εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 309. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην batch 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 310. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 311. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. μπάτζε 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 312. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 314, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε από κοινού την τροπολογία 314, λήξη, απορρίπτεται. ...314 και badge 8 άρχεται λήξη απορρίπτεται Τροπολογία 315 άρχεται πέρας εγκρίνεται πάμε στην 316 άρχεται πέρας εγκρίνεται Πάμε στην 319. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στις αιτιολογικές ε, σκέψεις. Τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 49. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 2, έναρξη. Πέρας, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 3, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 52, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 54 τροπολογία τώρα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην Τροπολογία 57 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τώρα άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 59. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 60. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 62. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 60, 63 Τροπολογία 63. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6α. Άρχεται. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 70 η 86 άρχεται. Πέρας. Για 10. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η 88 άρχεται. Ε, απορρίπτεται. Η 92 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 12 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 93 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 94 Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 99. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 100. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν τώρα στην τροπολογία 101, άρχεται, πέρας, απορρίπτεται, η 102 άρχεται, πέρας, εγκρίνεται, 103 και 104 ταυτόσημες άρχεται, Πέρας. Εγκρίνεται. 105. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 106. Πέρας. Απορρίπτεται. 107. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 198. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 109. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 14. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 111. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην τροπολογία 112. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 113. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 15. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 114. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 115 και 116 ταυτόσημες άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Και ε, τώρα η τελευταία ονομαστική ψήφος άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για την απόφαση, για την έναρξη διαπραγματεύσεων, έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Επόμενο σημείο προς ψηφοφορία είναι για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, για συνεργατικά έξυπνα συστήματα μεταφορών. συντάκτρια κυρία Γκραπίνη, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, μόνο να ψηφίσουμε. Ε, ωραία, ευχαριστώ. Ψηφίζουμε πρώτα τη συμβαστική τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Γκραπίνη, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι, μόνο να ψηφίσουμε. Ε, ωραία, ευχαριστώ. Ψηφίζουμε πρώτα τη συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 14. Όχι το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 14. Αυτό μου λένε εδώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 εγκρίνεται. Τροπολογία 18 στη συνέχεια. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορεί να η ψηφοφορία. Mm. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Mrs. Garcia. So we can continue. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι θέλετε να βγείτε από την αίθουσα, βγείτε. Όσοι θέλετε να μείνετε, μείνετε, αλλά καθίστε παρακαλώ. Για να συνεχίσουμε. Έχουμε μαζί μας την εισηγήτρια. για την ετήσια έκθεση 2016 για την προστασία των ε, οικονομικών συμφέροντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτης. Παρακαλώ καθίστε. Στι 27 Ιουλίου 2017 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά τη απάτης η ΟΛΑΦ δημοσίευσε την ετήσια έκταση για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφεροντών τη Ένωση και την καταπολέμηση κατά τη απάτης. Η έκταση καλύπτει τα μέτρα που πήρε η Επιτροπή για τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση τη απάτης και παρουσιάζει τα αποτελέσματα. Η Επιτροπή ελέγχου κυρίω για το ποινικό δίκαιο. Φέτος η κυρία Κουντρίτσκα είναι η εισηγήτρια για την γνωμοδότηση και θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης ε, σήμερα. Έχετε το λόγο κυρία Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα. και πρωτού ξεκινήσετε παρακαλώ να συνεχίσετε τις συζητήσεις εκτός της ευθύνης. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Κουντρίτσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για το σχέδιο έκτασης ε, του κ. Παρνιού της Επιτροπής Ελέγχων 17 και νομίζω ότι η γνωμοδότηση αυτή θα αποτελήσει μια ωφέλιμη συνεισφορά σε ό,τι αφορά και την τελευταία το τελικό σχέδιο του ψηφίσματος και αποτελεί και ένα σπουδαίο θέμα για συζήτηση. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία εγώ ως πιστεύω ότι είναι σημαντικά. Μία σύνδεση μεταξύ Eurojust, OLAF και EPPO, προκειμένου να μην υπάρχει ε, αλληλεπικάλυψη αρμοδιότητα. Σε ό,τι αφορά το, τις αρμοδιότητες του EPPO, ενδεχομένως να πείσουμε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν ήταν πρόθυμα για να μπορέσουμε και εμείς να διασφαλίσουμε αυτές τις, ε, αυτή την ανεξαρτησία. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να σας Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταμάτησε τη δημοσίευση τη ετήσια έκθεση για την διαφθορά μα. Είχαν υποσχεθεί κάθε δύο χρόνια με τέτοια έκθεση. Πιστεύω ότι όλη η διαδικασία παρακολούθηση ε, τη διαφθορά ήταν αρκή. Πιστεύω ότι αυτό στέλνει λάθο μήνυμα σε όσου ότι ε, η δική μας εργασία επιδεινώνεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αυτές τις απάτες καρουσέλ, σε ό,τι αφορά διαφθορά σε επιχειρήσεις. Συνεχίζει να γυρίζει και υπονομεύει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Κάθε έτος αυτό κοστίζει στην Ένωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Κουντρίτσκα. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κινίτση που είναι ασκιωδής εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ και τη συνάδελφο την κυρία Κουντρίτσκα για τη δέσμευσή της ε, για την ε, διατήρηση ε, της γνωμοδότησης λίγο για να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο για τα πραγματικά κρίσιμα σημεία για την κατεπολέμηση της απάτης και τις ζημίες των εισφορέων των χωρών. Ε, το κείμενο αποτελεί πολύ καλό εφαλτήριο που αντιπροσωπεύει και κρίσιμα ε, στοιχεία των ΠΙΦ ε, και τον κανονισμό ο οποίος συστηνεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επιτέλους δηλαδή η Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ποινική νομοθεσία για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφορών της Ένωσης. Και για πρώτη φορά θα υπάρχουμε και, και σημαντική αυτή η διαδικασία αυτή τη στιγμή βεβαίω ελπίζουμε το νέο κεκτημένο να τεθεί σύντομα σε ισχύ. Ε, Δυστυχώ για άλλη μια φορά εκρεμεί αυτή η πικρία το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δεν ε, ε, είχε ομοφωνία μεταξύ όλων των χωρών. Στήσω την κυρία Κουντρίτσκα πραγματικά πάρα πολύ διότι και τώρα επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να συσταθεί το συντομότερο Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να υπάρχουν σαφείς κανόνες για τις σχέσεις με τις άλλες υπηρεσίες, με την Όλαφ και φυσικά και τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά των συμφερόντων της Ένωσης. Τα περισσότερα πράγματα εξαρτώνται από την καλή συνεργασία μεταξύ των οργάνων της Ένωσης και επομένως πρέπει να υπάρχει μια βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων και κοινή δουλειά. Πιστεύω λοιπόν ότι εμείς σήμερα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο διαθέτουμε τα εργαλεία για να μπορέσουμε πραγματικά να εργασία μεταξύ συναδέλφων και βεβαίως ε, ε, η Επιτροπή μας θα μπορεί μέσω αυτής της δουλειάς ε, την οποία θα προσπαθήσω και εγώ να βοηθήσω μέσω κάποιων τροπολογιών να μπορέσουμε να δώσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού περισσότερα στοιχεία για να εμβαθύνουν και να μπορέσουν να εξετάσουν τις εργασίες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καλώς ορίζω το σχέδιο έκθεσης ε, της εισηγήτριας. Πάντα υποστηρίζα την ε, οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφέροντων της Ένωσης και ήμουν και υπεύθυνη ε, για την κατάρτιση της έκθεσης για τον ΕΠΠΟ. Είναι πολύ αποτελεσματική στην καταπολέμηση της απάτης, τη απάτη καρούς, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Ελπίζω λοιπόν η οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση, η οδηγία ΠΥΦ, να καλύψει και το ΦΠΑ το 10 εκατομμυρίων ευρώ είναι υπερβολικά υψηλό. Ελπίζω να το μειώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την πρώτη τη αναβρία συνένεση με του συζητητέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Λόπος προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα την ξεκίνησε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η Σεσίλια Γουάλστρομ ουσιαστικά ε, ε και δικαστική συνεργασία, ευθυγράμμιση ε, με την εθνική νομοθεσία, την καλύτερη δυνατή δικαστική συνεργασία και επιτέλους ευρωπαϊκή μέτρα για τα τεράστια ποσά τα οποία εμπλέκονται, τα οποία αφορούν όχι μόνο τη διαφυγή από τα φορολογικά στις νεότερες γενιές και για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα το οποίο δημιουργήθηκε λόγω της διαφθοράς και να συνεχούν ε, με το δικό τους τρόπο. Και νομίζω ότι εδώ από την ε, ερευνητική. Υπάρχει περιθέριο ευοληξίας για να μπορούν να συγκαλύψουν ε, απάτη, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Γι' αυτό ακριβώ και θα πρέπει να... Of ε, να διαβρύνει και αυτή την ενισχυμένη συνεργασία η οποία ξεκίνησε συμπεριλαμβανομένων και των ε, στοιχείων που ακόμα ε, περιμένουμε. Δηλαδή την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαίου Ισαγγελένα και συγκεκριμένων εργαλείων που θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να συνεργαστεί με τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και τους δημοσίους εισαγγελείς των κρατών